Αποχές εγκρίνεται λοιπόν το ψήφισμα. Φτάσαμε και στο τέλος των ψηφοφοριών. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι το ΕΛΚ ζήτησε ο κύριος Γκέρι να γίνει μέλος της ειδική Επιτροπής για την Οικονομική Κρίση. Νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε αυτόν τον διορισμό. Ο κύριος Πόσελ ζητάει το λόγο. Διαδικαστικό. Ζητώ συγγνώμη, αλλά σήμερα όλη την ημέρα έμαθα ότι μία ακροαριστερά από την Ουγγαρία κάθε φορά που παίρνει το λόγο μιλάει για την Ουγγαρία. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουμε ημερήσια διάταξη και κάποια θέματα που τα συζητάμε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Δεν είναι παρούσα όμως η συνάδελφος, αλλά νομίζω ότι θα ενημερωθεί. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα σας υποβληθούν την επόμενη συνεδρίασή μας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να διακόψουμε την συνεδρία. Σας εύχομαι όλους καλό ταξίδι.